ευρωπαϊκών πολιτικών όπως και άλλες περιφέρειες στον Ηνωμένου έχει πραγματικά μετασχηματιστεί. Ε, εδώ ολοκληρώνεται στις 8.30 αύριο το πρωί. Θα